Ξεκινάμε λίγο καθυστερημένα, αλλά είχαμε πολλή δουλειά κατά τη διάρκεια του γεύματος. Ξαναρχίζουμε τη συνεδρίαση τη επιτροπή. Πέρασε δυομίση ούτως ή άλλως. Νομίζω το πρωί την εγκρίναμε την ημερήσια διάταξη. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη. Πρώτο θέμα για την μερίσια διάταξη για το απόγευμα είναι το άρθρο 43 επικουρικότητα. Um. Um, so we have Υπάρχει μια αιτιολογημένη γνώμη από τα Εθνικά Κοινοβούλια που θέλει να ανακοινώσουμε, που να ανακοινώσουμε στην Ομαδική Ευώς. Ζητώ συγγνώμη ε, για την ενόχληση πρωτού περάσουμε στο σημείο της μερίσιας διαταξής. Θα ήθελα να επισημάνω το εξή. Θα ήθελα να επισημάνω το εξή στους συναδέλφους, λοιπόν. Ο κύριος Τροσάνη ε, αντικαθιστά τον κύριο Σάιερ στην ε, ψηφοφορία. Αν έχετε λοιπόν προσωπικές ερωτήσεις, ε, μπορείτε να τις θέσετε διμερώς. Αν υπάρχουν φυσικό ερωτήσεις. Όχι στην συναντρίαση, εκτός ημερήσιας διαταξής, αν το επιθυμείτε. Αυτό ως προσφορά προς τους ε, συμμετέχοντες. Μάλιστα. Ωραία. Το καταγράφουμε και συνεχίζουμε τη διάταξη. Τα διάφορα είναι για αύριο. Για αυτό το θέμα θέλετε, νομίζω καλύτερα να συνεχίσουμε με τη συνάντηση. Να σας διαβάσω την αιτιολογημένη ναι, γνώμη ή το έχετε δει το αναγγείλω στην ομάδα. Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών συστημάτων ενημέρωσης στον τομέα της ε, αστυνομικής συνεργασίας του ασύλου και της μετανάστευσης και ε, τροποποιεί τον κανονισμό της Eurodac. Η γνώμη είναι, ε, αφορά την πρόθεση της υλοποίησης των διευρωπαϊκών... Ε, το δεύτερο, η δεύτερη είναι η πρόθεση της υλοποίησης των ε, διευρωπαϊκών δικτύων. 5. Έτοιμα από το ΦΕΙΤΑΣ, από τη ΦΑΝΤΕΣ, είναι η Ισπανική Ένωση Ανάδοχων Οικογενειών, για ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Ο κύριος να μιλήσει. Ε, έγινε λάθος γιατί είπαν στη διερμηνία ότι ήμουν εγώ εισηγητής, αλλά δεν είμαι εγώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εξ ονόματος ε, της ομάδας ECR για την πρόταση της εισηγήτριας ε, και τη λύση που υιοθετείτε γιατί σε σχέση με την αναφορά που σχετίζεται με αυτή την ένωση υπάρχει ε, κάτι λάθος. Και πάλι ευχαριστώ την εισηγητρία γιατί τα θέματα ε, της εθνικότητας και του αστικού δικαίου είναι αρμοδιότητα κρατών μελών η κατάσταση στην οποία μπορεί να βρίσκονται οι ανήλικοι που προέρχονται από ρουμανικές οικογένειες ε, στην Ισπανία να καταλήξουν απάτριδες ε, δεν είναι ευθύνη του Ισπανικού κράτους αλλά του Ρουμανικού κράτους που δεν τους επιτρέπει να διαβιβάζεται η υπηκότητα στην περίπτωση αυτή. Και τρίτον, ε, η Ισπανική νομοθεσία λέει το εξή. Ρυθμίζεται στην Ισπανία, όλα, ρυθμίζονται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα των αλλοδαπών στην Ισπανία και ε, εγγυώνται για στην Ισπανία υπάρχει η εγγύηση της ελευθερίας ε, μετακίνησης ε, και υπάρχει η συμμετοχήριση και των ολοδαπών και των ημεδαπών και οι ελοδαποί που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και στη βασική κοινωνική πρόνοια. Γι' αυτό Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την επιστολή της και την πρόταση, γιατί κατανοώ ότι πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμία παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανηλίκων και μάλιστα επιπρόσθετα βάσει της ισπανικής νομοθεσίας αναγνωρίζεται η δυνατότητα να αποκτήσουν την ισπανική υπηκότητα όταν ε, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ευχαριστώ. Thank you. Does any other member wish to comment on this? Κάποιος άλλος θέλει να σχολιάσει την ε, αναφορά αυτή. Η Κομισιόν. Όχι. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ της επιστολής. Ψηφίζεται ναι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σημείο 6. Δεν έχουμε τίποτα.